Δικό σα φταίξιμο ενάν η Ευρώπη όλο και λιγότερο αρέσει. Έχετε κλειστεί στου πύργου σα και δεν μπορείτε να εισακούσετε και να απαντήσετε στι απαιτήσει προσδοκίε των πολιτών. Ε, ε, πηγαίνετε κατά των λαϊκιστών, γιατί δεν μπορώ να δώσετε απαντήσει στο λαό. Αλλά πρέπει να πω πραγματικά, συνεχίστε έτσι. Ε, μην κάνετε αυτοκριτική και α εφευρίσκετε πάντα δικαιολογίε συνωμοσιακέ για τη λαϊκή ψήφο. Εμεί θα εξακολουθούμε να απαντούμε στις προσδοκίες των πολιτών και θα προστατεύουμε τα συμφέροντα της χώρας μας με υπερηφάνεια και με υψηλά το κεφάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο Σνάρφος Γκραζοντέψκι για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά έχουμε συζήτηση για το ίδιο θέμα. Το θέμα μοιάζει να είναι πολύ σημαντικό, όμως ε, η συζήτηση ίσως να μην ήταν και απολύτως απαραίτητη. Έχω την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πέσει στην παγίδα της ε, συνωμοσιολογίας ε, γιατί πάρα πολλοί μιλάνε για παρεμβολή στις και παρεμβάσεις στις εκλογές, ενώ κατ' ουσίαν θα πρέπει να συζητάμε για παρεμβάσεις στις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρώπη. Παραδείγματο χάν ρωσική επιρροή στην γερμανική S5. Για δέστε τον Gerhard Schröder ή την Gazprom, το ρόλο που παίζει στη Γερμανία. Μετά μιλάμε για την Αυστρία και για την ε, ρωσική επιρροή μέσω του κυρίου Στάχερ και ε, επιρροή επίσης ε, προς τον πρόεδρο Μακρόν. Αυτό το διαπιστώσαμε ε, κυρίως σε αυτά που είπε ο κύριος Μακρόν στον Economist. Αυτά είναι πολύ σημαντικά προβλήματα και ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε και γι' αυτά. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Τσαρτσαλέχος ε, για δύο λεπτά παρακαλώ. Eh, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια κυρία Επίτροπε για την ε, επανεκλογή σας. Η παρέμβαση είναι γεγονός. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια στρατηγική. Γι' αυτό πρόκειται για ένα σχέδιο με συγκεκριμένο στόχο. Στόχος είναι να αποδυναμωθούν τα δημοκρατικά μας συστήματα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχουν λοιπόν να αποδυναμώσουν το δημοκρατικό σύστημα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και χρησιμοποιούν στο, αυτούς που στο παρελθόν κατέστρεψαν τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά συστήματα και την Ευρώπη. Τον εθνικισμό δηλαδή και τον λαϊκισμό. Ευτυχώς ε, ζούμε σε δημοκρατικά συστήματα και σε μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ε, επιτρέπεται να ακούγονται όλα τα παράξενα όπως ας πούμε ότι η Ομοσπονδιακή Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ είναι η ίδια εξωτερική παρέμβαση στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οι χώρες που προκαλούν, όπως η Ρωσία, η Κίνα και άλλοι, είναι υπαρξιακές προκλήσεις ε, οι παρεμβάσεις ε, αυτές δεν είναι μόνο μέσω των κοινωνικών δικτύων, είναι η χειραγώγηση των δικτύων, είναι διείσδυση ανθρώπων, είναι παραχάραξη ε, εγγράφων, είναι η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, αλλά και η στήριξη των οργανώσεων βιτρίνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εντοπίσει ενεργούς πράκτορες, κατασκόπους ε, του Ρωσικού στρατού και τελευταία υπόθεση ήταν ακριβώς στην Ισπανία όπου ερευνήθηκε η δραστηριότητα τέτοιων πρακτόρων στην Καταλωνία στην ε, εποχή Τη παράνομη ψηφοφορία του Οκτωβρίου 2017. Αυτή η απειλή δίνει νέο νόημα στην αποστολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω ε, θεματοφύλακα των συνθήκων. Αυτή τη στιγμή αποτελεί και τον θεματοφύλακα τη Δημοκρατική Αρχιτεκτονική τη Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε σαφεί στην καταγγελία, να είμαστε δραστήριοι στη χρήση όλων των μέσων, αλλά και να είμαστε σαφεί και να απαιτήσουμε ότι όλοι οι φορεί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, θα αναλαμβάνουν τι ευθύνε του στη στιγμή που πρέπει να δοθεί απάντηση σε αυτή την την απειλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Πίκουλα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι το θέμα αυτό επανέρχεται στην ημερήσια διάταξη ε, παρότι πρόσφατα απορρίφθηκε μια πρωτοβουλία των σοσιαλδημοκρατών. Εμείς ε, θέλαμε να συστήσουμε μια επιτροπή. Ε, διαπιστώσαμε στις πιο τελευταίες εκλογές σε διάφορες χώρες ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα της παρέμβασης κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες δημοσιεύουν διάφορα στοιχεία χωρίς έλεγχο έλεγχο. Οι πολίτε βέβαια έχουν εντοπίσει αυτό το πρόβλημα. Τα δύο τρίτα των πολιτών δείχνουν ότι ανησυχούν. Όμως όσον αφορά στις εκλογικές μας ε, διαδικασίες ε, δεν θα πρέπει να περιζόμαστε μόνο στη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Θα πρέπει να εξετάσουμε και την παράνομη χρηματοδότηση των κομμάτων. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι για άλλη μια φορά στους συναδέλφους να προβλέψουν μια εξεταστική επιτροπή που να εξετάσει την ε, ανάμειξη στις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Γιατί εδώ πρόκειται για την ε, προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Εκ τούτου οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις. Επόμενη, η συνάδελφος κυρία Γκίψον ένα λεπτό παρακαλώ. Εξετάζοντας αυτό το θέμα, θέλω να σας πω, αισθάνομαι σαν να έκανα μια φοβερή ανακάλυψη ε, σε ένα έργο του James Bond. Όλα μοιάζουν να οδηγούν στον Steve Bannon, η σκευωρία οδηγεί στον Steve Bannon, ο οποίος ομολόγησε ότι θέλει να χρηματοδοτήσει ένα εθνικιστικό κίνημα για να αναλάβει ταινία του κόσμου. Αυτή η σκευωρία είναι απίστευτη γιατί αυτός είναι πίσω από την Cambridge Analytica. Ε, αυτό η, μια μηχανή η οποία, συν, η οποία ταυτίζεται με σκοτεινό χρήμα, με ψευδές ειδήσει, με στόχο να αποθανηθούν οι άνθρωποι να ψηφίσουν. Τα στοιχεία είναι σημαντικά δείχνουν ότι όλα αυτά επηρέασαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο του Ηνωμένου Βασίλειου. Ο Μπέραν είναι μαριονέτα, πίσω από αυτόν είναι ο Φαράζ, ο Τραμπ. Οι έρευνε έχουν αποκαλύψει ε, μαύρο χρήμα που διοχετεύθηκε στι προεκλογικέ εκστρατείε. Πρόκειται για μια στρατηγική εκστρατεία ε, που απειλεί όχι μόνο το αποτέλεσμα εκλογών, αλλά και τι δημοκρατίε μα και τι ελευθερίε μα. Και όλα αυτά πρέπει να αναχαιτιστούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, συνάδελφος Τσάουνς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σήμερα συζητούμε την παρέμβαση από άλλες χώρες στις δημοκρατίες μας και στις εκλογές μας. Ένα θέμα το οποίο δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι είχαμε αρκετά ψέματα και παραπληροφόρηση. Λοιπόν, η ομιλία μου απαρτίζεται από τρία γεγονότα, στοιχεία και μία ερώτηση. Πρώτο στοιχείο. Στι 17 Οκτωβρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι μυστικέ υπηρεσίε και η Επιτροπή του Κοινοβουλίου μα ε, τελείωσε την έκθεσή τη για ρωσική παρέμβαση στι εκλογέ του Ηνωμένου Βασίλειου, κυρίω για τον Ιούνιο του 2016, το δημοσίφισμα για το Brexit και το υπέβαλε στην Downing Street. Έπρεπε να έχει δημοσιευτεί σε 10 μέρε, σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Ανατολική Επιτροπή, αυτή η έκθεση. Δεύτερον, είχαμε κάποιε διαρροέ από αυτή την έκθεση και βρήκαμε ότι η Ρωσία πράγματι μπορούσε να είχε επηρεάσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο και επίση θέτει ερωτηματικά η διασυνδέση μεταξύ Μπόρι Τζόνσον, που είναι ο παρόν πρωθυπουργό μα, με το Συντηρητικό Κόμμα και του Ρώσου δωρητέ. Τρίτο στοιχείο. Αυτό ο ίδιο ο Μπόρι Τζόνσον ε, αρνείται να δημοσιεύσει αυτή την έκθεση, την κατάσταση στα χέρια του. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ότι Ο πρόεδρο, ο Ντόμινγκ Γκριπ, πρόεδρο τη Επιτροπή, θεωρεί ότι αυτή ε, μα αποστομώνει. Μένει το στόμα ανοιχτό όσον αφορά ε, το ότι δεν δίνει την έκθεση δημοσίευση. Λοιπόν, με τέτοια απελπισία είναι η ερώτησή μου τι κρύβει ο Μπόρι Τζόνσον. Δεν πρέπει να είσαι ο Σέρλοκ Χόλμ για να φτάσει διαπαγωγή στο συμπέρασμα. Ευχαριστώ. Επόμενο, συνάδελφο Λαπόρτ, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ασχολούμαστε με το θέμα της εξωτερικής παρέμβασης στις εκλογές μας, θα βλέπουμε στην αυγή μπροστά μας η Ρωσία. Έχουμε μανία που θα δικαιολογούσε και κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και προσέγγιση ε, σαν να συμμετέχουμε στον ψυχρό πόλεμο που υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει μια παρέμβαση. Λοιπόν, θα έπρεπε να ε, θέλαμε ε, να ε, καταδικάσουμε την κυβέρνηση, επιβάλλουμε κυρώσει στον Ορμπάν γιατί παραβίασε του ε, κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και για του μετανάστε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε τον Ζω Όρο που έχει ΜΚΟ και προωθεί τη μαζική μετανάστευση και εξυπηρετεί τα πολιτικά συμφέροντα αντίθετα από τι σχέσει μα ε, που θέλουμε να έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, με την Βρετανική κυβέρνηση ε, θέλουμε να, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάσει. Το 2015 δημιουργήθηκε και μια task force που ήθελε να ελέγξει τις πληροφορίες που είναι αφισβητήσιμες, που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο για, το, για, για προβλήματα άλλα. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραπληροφόρηση συνεχώς που αναφέρουμε, μήπως είναι παραπληροφόρηση που δεν προσέχεται στα πλαίσια της ε, πολιτικής που ακολουθείτε. Τίθεται το ερώτημα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν για μία ακόμη φορά αφορά την παρέμβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο τους δεν είναι ε, παράμενο αδρανοί και θα έχουν κάποια νομιμότητα να συζητούν αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που λέτε ε, μεταφράζονται, ε. γίνεται διερμηνία. Ε, για φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει με την ταχύτητα που μιλάτε. Ευχαριστώ η παρέμβαση των ξένων χωρών στις εκλογικές διαδικασίες στην Ευρώπη είτε σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο δεν είναι κάτι καινούριο. Οι ξένες δυνάμεις πάντα προσπαθούσαν να ασκούν πολιτική επιρροή ε, επί των ευρωπαϊκών χωρών. Μεταξύ άλλων ε, χρησιμοποιούν και αυτό το μέσο με, λόγω τεχνολογίας είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι κατά παρελθόν. Η πρόθεση παραμένει η ίδια. Είναι σημαντικό να προστατευόμαστε από ξένε επιρροές όσον αφορά τι πολιτικές και άλλε διαδικασίε μας. Αυτό είναι προ όφελο των πολιτών μας. Είναι πολύ συχνά στόχο προπανδιστικών δραστηριοτήτων που έχουν στόχο να του παραπλανήσουν. Επίσης είναι σημαντικό να σταματήσουμε να αυταπατώμεθα ε, δικαιολογώντας μέσω άλλων τις αποτυχίες μας. Η αυξανόμενη απογοήτευση κατά της πολιτικής ελίτ και των δημοκρατικών θεσμών στην Ευρώπη όνο, μόνο εν μέρει οφείλεται στην ξένη προπαγάνδα. Επίσης οφείλεται και στην κακή δουλειά των Ευρωπαίων πολιτικών που είναι απόμακροι από τους λαούς. Ευχαριστώ. Ζούμε σε μια εποχή παραπλανητικής ενημέρωσης και όπως ε, το περιέγραψε η Λίδια Πόλγκριν, ε, Εξαπλώνεται ως ιός ε, η παραπλανητική ενημέρωση στο οικοσύστημά μας. Το πρώτο τρίμηνο του 2019, 2,2 ε, δισεκατομμύρια ψευδείς λογαριασμοί ε, ε, αφαιρέθηκαν από το δημοψήφισμα για το Brexit με τις εκλογές του Προέδρου Τραμπ μέχρι τις πρόσφατες σε παντού όλα αυτά επηρεάστηκαν από ξένες δυνάμεις. Επίσης Υπάρχουν ε, ειδικοί των μίντια ε, που αναζητούν την αλήθεια. Η συνένεση δεν είναι αλήθεια, η φήμη δεν είναι γεγονός, η καταστροφή των σταδιοδρομιών δεν είναι μεταρρύθμιση. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση. Πρόσφατα δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως τα ψευδή, οι ψευδείς ειδήσει είναι απειλή για τη δημοκρατία μας. Είναι ανάγκη να κάνουμε κάτι. Το να μην κάνουμε τίποτα θα υποσκάψει τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα ψεύδη ε, στο ίντερνετ. Δεν μπορεί να λειτουργεί το ίντερνετ όσο η άγρια δύση. Πρέπει να έχουμε κυβερνοασφάλεια, συστήματα τα οποία θα μπορούν να σταθούν να εντοπίζουν τις ψευδείς ειδήσει και την ξένες παρεμβάσεις. Με συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς σωστές πληροφορίες και στοιχεία, οι μοί μας δεν έχουν αξία και οι πολίτες μας δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας. Ε, θα πρέπει λοιπόν η ψηλότερη αξία να είναι η αλήθεια και τα στοιχεία. Ο κύριος Λόμπες Αγγιλάρ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο. Επίτροπε Γιουρόβα, συγχαρητήρια. Πολλοί από εμά με μεγάλη πλειοψηφία σα στηρίξαμε ε, για να εκλεγείτε και πάλι αντιπρόεδρος. Έχετε δικούς σας πόρους και θα ελπίζουμε πως θα αποκαταστήσετε την κοινωνική ατζέντα αλλά κυρίως την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών για τις οποίες είστε υπεύθυνοι. Ε, ε, σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης μιλήσαμε για πάλι για νέα επεισόδια παρέμβασης στις προεκλογικές διαδικασίες. Δεν γίνεται να μην αναφέρω αυτό που ξεκίνησε, την έρευνα που ξεκίνησε λόγω της παρέμβασης ενός ειδικού ρωσικού επιτελείου ε, κατασκόπων ε, στις ε, στο ισπανικό δημοψήφισμα Όλα αυτά γίνονται πάντοτε υπέρ του λαοκισμού, της ακροδεξιάς, του αντιδραστικού εθνικισμού. ούτε και με την Ειδική Επιτροπή που ζητήσαμε να συσταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο να φτιάξουμε μία δομή ευρωπαϊκής κατασκοπής που θα υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τίποτα δεν έχει περισσότερη αξία. Ευχαριστώ. Πίσω από το διάφορα άρθρα ε, που, λέει, λέει, που, που κυκλοφορούν στον τύπο λένε ότι η Ουγγαρία δεν θέλει τους μετανάστες. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μια ευρωπαϊκή απικία. Κάποια παραδείγματα παραπληροφόρησης ε, από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Περίπτωση που δεν έχετε παρατηρήσει, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Αγωνιζόμαστε για την αλήθεια. Όχι τη δική μας, όχι τη δική τους ε, αγώνας για αντικειμενικά στοιχεία και πραγματικότητα και χάνουμε. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα στοιχεία και τα ψέματα είναι ανακατεμένα. Ε, όμως πιστεύω πως έχουμε πολλά να προστατεύσουμε. Τα θεμέλια της δημοκρατίας μας εξαρτώνται από την ικανότητά μας να υπερασπιστούμε τις αξίες μας και τις αρχές μας ε, και την αντικειμενική αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινότητα κοινών αξιών θα πρέπει να είναι στο μέτωπο αυτού του αγώνα. Το Brexit ήδη διαπιστώσαμε πώς αυτή η παραπληροφόρηση οδηγεί σε αποσύνθεση και για μια φορά η ιστορία δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Το ρόλο λοιπόν, το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κρά για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ μεγάλωσα στο κομμουνιστικό κομμάτι της Γερμανίας και θυμάμαι τα σχολικά βιβλία όπου ανέφεραν ότι το ΡΙΑΣ, ο σταθμός στο Βερολίνο ή το Free Europe ε, προσπαθούσαν να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες ε, στη δική μας τη χώρα. Και γι' αυτό λοιπόν, ακούγοντας όλες αυτές τις ε, συνωμοσιολογικές θεωρίες του αδέλφου Γκίψον και την ισπανική πρόταση που λέει να, υπάρχει μια, να υπάρχουν ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι επιλέγουν ε, κόμματα ε, που τους αρέσει η πολιτική και καταψηφίζουν άλλα που δεν τους αρέσει η πολιτική τους. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι και από τους ιδιωτικούς σταθμούς και από τους δημόσιους δεν μπορούν να ενημερωθούν επαρκούς. Γιατί σε έναν κρατικό σταθμό ποιος μπορούσε να εξηγήσει γιατί εξελέγει ο Τραμπ. Εκεί αναφέρονται μόνο συνωμοσιολογίες αλλά καμία ενδελεχής ανάλυση. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για τη δημοκρατία θα πρέπει να αντέχει τον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα των απόψεων. Ε, δεν είναι δυνατόν όμως με μυστικές υπηρεσίε, να προσπαθήσει κανείς να φημώσει τους άλλου που δεν, τους αρέσει, δεν του αρέσει η άποψή του. Ο στάδιος κ. Τσανέτσκι για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ε, είναι ε, η πρώτη σας εμφάνιση εδώ μετά τις εκλογές. Και για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια ψήφισα για σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να πω λοιπόν το εξής. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά ε, για το θέμα αυτό, αλλά δεν πρέπει βέβαια και να το δαιμονοποιούμε. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αλλά επίσης ε, δεν είναι ιδιαίτερα ωραίο αν εκείνοι που χάνουν τις εκλογές αποδίδουν την ήττα τους ε, σε εξωτερική παρέμβαση. Δεν είναι σωστό αυτό. Ε, θα πρέπει λοιπόν να σας προειδοποιήσω να μην είμαστε μονόπλευροι όταν εξετάζουμε την κατάσταση. Γιατί όταν ακούω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη Ρωσία και ότι υπάρχει μόνο ο Στίβ Bannon, έχω την εντύπωση ότι αυτοί που το λένε ζουν σε έναν εικονικό κόσμο. Ε, για ελάτε να δείτε λιγάκι την πραγματικότητα. Όχι μόνο η Ρωσία και άλλοι βέβαια ανακατεύονται και γι' αυτό πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Επόμενο συνάδελφο, ο κ. Αρλούκοβιτ για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, ζούμε ε, σε ενδιαφέρουσες αλλά δύσκολες εποχές. Ζούμε σε εποχές ε, όπου για να επιτύχει κανείς αποσταθεροποίηση δεν επιτίθεται με τάγκ ή με υποβρύχια. Σε αυτές τις ενδιαφέρουσες εποχές που ζούμε θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε την ευθύνη που φέρουν οι πολιτικοί. Εγώ είμαι γιατρός. Η ιατρική λοιπόν μου έμαθε ότι καταρχήν το πρόβλημα για να το λύσει κανείς πρέπει να το αναλύσει και μετά να κάνει μια σωστή ε, διάγνωση. Εδώ πρόκειται για την ε, ασφάλεια των παιδιών μας. Αυτή μας έχει ανατεθεί. Αν λοιπόν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αν συνειδητοποιήσουμε ότι για τις μεγάλες δυνάμεις αυτό που τις ενδιαφέρει είναι να αποσταθεροποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τότε δεν μπορούμε να τους ανοίγουμε διάπλατα τις ε, πόρτες. Για δέστε λιγάκι την ε, στρατική Γερασίμοφ. Ήταν ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων στη Ρωσία και είχε γράψει σε 7 σημεία τι πρέπει να γίνει για να αποσταθεροποιηθεί ένα κράτος χωρίς ούτε καν να χρησιμοποιηθούν τα τάγκς το πρώτο σημείο, αποσύνθεση της κοινωνίας. Άρα δηλαδή να ε, διχαστεί η κοινωνία, να τσακώνονται οι κοινωνικές ομάδες μεταξύ τους. Το δεύτερο που έγραψε ήταν η υποβάθμιση των ελίτ. Αυτό δηλαδή σημαίνει ε, να υποβαθμιστούν οι ελίτ για να είναι πιο εύκολη η χειραγώγηση των ε, πολιτών. Τρίτον, αποσύνθεση και επίθεση στις διοικήσεις των κρατών. Διερωτώ μετά, δεν συμβαίνει αυτό σήμερα. Τέταρτο σημείο, συγκεντρωτισμός και συγκέντρωση της εξουσίας. Και εδώ και σε εμά πρέπει να δούμε μήπως υπάρχει συγκεντρωτισμός. Και τέλος, αλλαγή της ιστορίας, αλλαγή των ε, ηρών και το τελευταίο το σημείο, καταστροφή του δικαίου. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να διερωτηθούμε, ο Γερασίμοφ έχει προβλέψει πολύ καλά το πώς μπορούν να αποσταθεροποιηθούν τα κράτη. Επόμενος ε, ομιλητής. Για ένα λεπτό, ο ε, κύριος ε, Ο κύριος Ζωγίνιο. Είμαστε μια παγκόσμια αναφορά όσον αφορά την κράτος δικαίου, την ελευθερία και την ε, πολιτική επιλογή. Αυτή τη στιγμή όμως όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε ε, πολύ έντονη παρέμβαση, πληροφορίες άπλετες, ε, αληθείς ή ψευδείς και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια γενική, ένα γενικό αγώνα. Και τι άοπλα έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε γενικά την ε, εκπαίδευση την ψηφιακή και την καθολική πρόσβαση στο ίντερνετ. Η εφαρμογή των κοινών αξιών, η εμβάθυνση ενός εσωτερικού κώδικα διοντολογίας που περιλαμβάνει και τις ε, ε, διεθνείς εταιρικέ σχέσεις έχει νόημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπερασπιστούμε τη την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και κάθε πολίτης να είναι ένας στρατιώτης αυτόν τον αγώνα, γιατί οι υπόλοιποι συνεχίζουν να προσλαμβάνουν για να μας αποδυναμώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για, για υπευθυνότητα. Έχουμε τις ευθύνες εκείνων που ε, να υπερασπιστούμε τους πολίτες έναν της παραπληροφόρησης. Πρέπει να τα πούμε ότι πρόκειται περί ασύμετρης επίθεσης και είναι υπεύθυνη η Ρωσία και η απάντησή μας η πολιτική πρέπει να είναι στο ύψος της επίθεσης. Μετά είναι και ευθύνη εκείνο που διαχειρίζονται την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για αυτή την ε, ε, επίθεση. Μεγάλες πλατφόρμες που, είναι, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και δίνουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο δεν έχουν επαρκή ασφάλεια. Θα πρέπει να γίνει σωστή ανάλυση και αξιολόγηση και θα πρέπει οι πλατφόρμες να είναι πιο διαφανείς και να δείξουν ότι είναι πραγματικά υπεύθυνες. Εν συνεχεία, αν πάρουμε σοβαρά τις απειλές κατά της δημοκρατίας, θα πρέπει να βρούμε τους αναγκαίους πόρους για να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα και θα πρέπει να συζητήσουμε με σοβαρότητα αυτές τις ευθύνες. Ευχαριστώ. Mm. Mm. Uh, Στο Πρόεδρε, πολύ σημαντικό το θέμα η παρέμβαση στην ευρωπαϊκή δημοκρατία στις εκλογές. Είναι άμεση παραβίαση της κυριαρχίας των κρατών μελών και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοια. Είναι βασικό όλα τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι συγκεκριμένα όσον αφορά τι κυβερναπηλέ ότι έχουν πολιτικέ ασφαλεία και που είναι αποτελεσματικέ και θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Όμω, η παρούσα τάση να ε, κατηγορούμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα εκλογών σε ξένη παρέμβαση πρέπει να σταματήσει. Η αριστερά ήταν διαβόητη να κατηγορεί για αυτό το θέμα ε, για αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα ότι γι' αυτό φταίνουν οι ξένε δυνάμει. Δεν υπονομεύουν έτσι την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία αλλά υποτομούν και την ευφία των Ευρωπαίων ψηφοφόρων. Εξίσου, ο αντίκτυπο τη διάδοση παραπληροφόρηση από ξένε δυνάμει και τοπικού φορεί, παρομοίω δεν πρέπει να υποεκτιμηθεί, να υποτιμάται. Πρέπει να πούμε ότι δεξιά, ακροδεξιά κόμματα δυσανάλογα και άδικα κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποίησαν και επωφελήθηκαν από τέτοια παραπληροφόρηση. Σχετικά με αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι κάθε μορφή παραπληροφόρησης θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Ακόμα σύμφωνα με, τις, ε, με ισότητα κάτω δικαίου και δημοκρατία και όταν απευθύνεται κατά δεξιών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία ή ο κύριος Σόφρα. Monsieur Président, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή τη συζήτηση δεν θέλουμε να εμποδίσουμε του ηγέτε κάποιου ξένου χώρα να εκφράσουν το όραμά του για τον κόσμο τι προτιμήσει του. Θυμόμαστε ότι ο Φρανσουά Ολόν ε, ε, ε, την, την πρόεδρο τον είπα το 2016 είχε εκφράσει προτίμηση και ένα χρόνο τώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στους Πολωνούς όχι χωρίς κάποια λαζονία να έχουν καλύτερους ηγέτες Στόχο τη συζήτηση δεν πρέπει να είναι να ευχόμεθα ότι οι πολιτικοί υπεύθυνοι δεν μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους. Το πραγματικό θέμα είναι αυτό τη φύσεω και των μέσων που χρησιμοποιούνται για να γίνει αυτό. Ε, σήμερα κάποιες ξένες δυνάμεις κατάλαβαν ότι πάνω από το μισό των Ευρωπαίων πληροφορούνται μόνο από τα κοινωνικά δίκτυα. Ενημερώνονται από εκεί και χάρη σε μια χρήση ε, ε, των ρομπότ και τεχνικής νοημοσύνης, ηλεκτρονικό ρομπότ, Πολλοί που βγαίνουν στο διαδίκτυο στην Ευρώπη δυστυχώς καταλήγουν να πιστεύουν ανωνύμους που ανεβάζουν δυσφημιστικές ειδήσει για τους, ε, για τους, ε, αυτούς που τους δικούν δημοκρατικά. Πάνω από 150.000 λογαριασμοί στα αγγλικά ήταν οι λογαριασμοί στο διαδίκτυο μερικές εβδομάδες πριν την ψηφοφορία για το Brexit και αυτό ούτως ώστε να αποσταθεροποιήσουν την Ευρώπη. Σας ανακοινώνω λοιπόν ότι τις επόμενες ημέρες θα ζητήσω από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τη συγχαίρω, ώστε να καταρτήσει ένα πρόγραμμα εντοπισμού των μηνυμάτων που προέρχονται από ξένες ε, δυνάμεις ούτω ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε στα κοινωνικά δίκτυα τον πληθυσμό όταν μάλιστα είναι προεκλογική περίοδος. Τα τεχνολογικά μέσα για αυτό τον φιλόδοξο στόχο υπάρχουν ε, και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να είναι πολύ πιο επιθετική και να ανταγωνιστεί τους, εκείνους που χειραγωγούν τις ειδήσει στο έδαφος τους. Δεν θα πρέπει να γίνουν υπηρέτε ψηφιακοί των ρωσικών αμερικανικών συμφερόντων εκείνοι που βγαίνουν, οι Ευρωπαίοι που βγαίνουν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, ο ολοκληρωτισμός είναι όταν η διάκριση μεταξύ γεγονότος και φαντασίας δεν υπάρχει πλέον κάποιος. Η αφέλεια της Ευρώπης δυστυχώς δεν είναι ε, κάτι φανταστικό, τουλάχιστον η αντίδραση όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας είναι ρεαλιστική, μια πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια, κύριε Επίτροπε, για την επανεκλογή σα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα. Από το 2015 η Ένωση δήλωσε ότι θα ε, ασχοληθεί ενεργά ε, δραστήρια με τις ψευδείς ε, ε, ειδήσει και την παραπληροφόρηση. Έγιναν εκλογές και στο ίμιση των χωρών του ΟΣΑ στη διάρκεια αυτών των προεκλογικών διαδικασιών υπήρξαν εξωτερικές παρεμβάσεις και ξέρουμε ότι ορισμένε ήταν στοχευμένες. Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις χώρες μας. Υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις online και παραποίηση πληροφοριών και αυτό αλλάζει τις γνώμες των των εκλογέων. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέπουμε να υπάρχουν αυτές οι αποκλήσεις από τους νόμους. Η δημοκρατία διέπεται από νόμους και υπάρχουν και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση. Δεν μπορεί κάθε κράτος να ρυθμίζει τις πληροφορίες που περνούν από τα σύνορα. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα projects για να καταπολεμήσουμε τα fake news και τις ε, ε, παρεμβάσεις σε κάθε χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρένα. Thank you. Η κυρία Φωνφίση Ειρήνα, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Γιούρεβα, παρά ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλης κλίμακας, ε, ότι υπήρξε μεγάλης κλίμακας ε, επιρροή από ξένες δυνάμεις στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016, δεν επαναλήφθηκε το δημοψήφισμα. Επίσης, οι ειδικοί είπαν ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλτ Τραμπ επηρέασαν αυτό το, ε, το δημοψήφισμα και οι, ήθελαν, και οι δύο ήθελαν να προάγουν το Brexit και να αποδυναμώσουν την Ένωση. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις εκλογικές μα νομοθεσίε και να βελτιώσουμε την εποπτεία των μέσων ε, μαζικής Ε, Παλαιότερα το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αποφασίσει περί νομοθεσίας. Ο Μπόρι Τζόνσον αγνόησε την ακυρεότητα της δημοκρατίας μας και το καθήκον του να προστατεύσει του πολίτε. Γιατί, γιατί αν ερευνούσε αυτό το ζωτική σημασία θέμα θα οδηγεί το σε δυο επιθυμητές ε, ε, ερωτήσεις ε, για το δημοψήφισμα. Γι' αυτό ο Μπόρις Τζόνσον απέφυγε να αποκαλύψει την έκθεση περί ρωσικής παρέμβασης. Καιρός είναι να ξεφορτωθούμε τον Μπόρις Τζόνσον και να δώσουμε στο βρετανικό λαό τη ζωή που αξίζει. Η κυρία Ματίλτε Αντρουέ. Αν και αυτή η συζήτηση ξεκίνησε για να κακολογήσουμε τη Ρωσία, εγώ θα αποκλίνω από αυτόν τον κανόνα για να, κατακρι... καταγγείλω την παρέμβαση της Τουρκίας που δεν κρύβει τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες και που δεν είναι καθόλου φιλικές. Οι πρόσφατε ε, τουρκικές γεωτρήσει στα ε, κυπριακά χωρικά ύδατα δεν κρύβουν τις ε, προθέσεις και επίσης το θέμα της κροή μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ποια είναι η στάση της χώρα αυτής. Όταν οι κάτω χώρες και η Γερμανία προσπάθησαν να κάνουν να καταστήλουν μάλλον ε, τις ε, απειλές του Ερντογάν. Αυτός καλεί τους ε, Τούρκους μετανάστες που ζουν στις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν πολλά παιδιά για να αλλάξουν τα πράγματα. Επίση, παρέμβαση όσον αφορά την ελευθεροτυπία. Όταν ο κύριο Ερντογάν επικρίνεται στις, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι άνδρες του επιτίθενται στα περίπτερα. Επίσης, όσον αφορά τα σχολεία, ο Τούρκος ε, υπουργό Εξωτερικών καταδικάζει την γαλλική γερουσία. Δυστυχώς δεν είναι όλα αυτά που έχει κάνει η Τουρκία, υπάρχουν και άλλα. Η Τουρκία λοιπόν καλά θα κάνει να βλέπει, να κοιτάει τι κάνει και να πάψει να παρασταίνει τον ε, Σουλτάνο ο Ερντογάν. Δεν πρόκειται εκείνο να γίνει ηγεμόνα τη Ευρώπη και θα πρέπει να του το θυμίσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπενχιουμέα Ιζαμπέλ. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η παρέμβαση ε, ξένων δυνάμεων ε, κάθε φορά επηρεάζει την ελευθερία που έχουμε για να εκλέγουμε τους, τους ε, αρχηγούς μας και τους ε, ε, πολιτικούς μας. Είναι μια από τις μεγαλύτερες μας ελευθερίες. Δεν μπορούμε παρά να πούμε πόσο ηρωικά οι Βάσκοι στην Ναβάρα για δεκαετίες υπερασπίστηκαν την ελευθερία ε, καταστέλλοντας το τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ και καταγγέλλοντας τον τρόμο που προκαλούσε για να μπορέσει έτσι να καταλάβει πολιτικό χώρο που δεν της ανήκε. Ο κύριος Περνάντο Βαρένα που έχει καταδικαστεί επειδή ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ σήμερα είναι ευρωβουλευτής ωστόσο. Υπάρχουν και εσωτερικές ε, όμως απειλές ε, που μπορεί να προκληθούν λόγω της αποτυχίας του πολιτικού μας, ε, της αποτυχίας του πολιτικού συστήματος. Οι παρεμβάσεις ε, γίνονται για να στηρίξουν ε, αυταρχικά καθεστώτα και λαϊκιστικά κόμματα. Είδαμε παρεμβάσεις στη διάρκεια του δημοψηφίσματος για το Brexit, για τις εκλογές τις γαλλικές και το ίδιο είδαμε στην Ισπανία στην κρίση την αποσχιστική της Καταλωνίας το 2016. Θα έχουμε διαρκώς επιθέσεις, πρέπει αυτό να το πάρουμε απόφαση, επιθέσεις κατά της σταθερότητά μας και άρα και της ελευθερίας μας. Ορισμένες επιθέσεις είναι προφανείς, άλλες αόρατες, αλλά ε, διαταράσουν ε, τις εξελίξεις. Ε, ο στόχος όλων αυτών είναι ο ίδιος, να μας αυστεροποιήσουν, να μας διχάσουν και τέλος να μας αποδυναμώσουν. Πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα, περισσότερες κοινέ πληροφορίες για να μπορέσουμε να χαιτήσουμε τα ανεπιθύμετα αποτελέσματα, περισσότερη ενότητα. χρειαζόμαστε τους θεσμούς που να αγγιώνται την καθαρότητα και την ανεξαρτησία των εκλογικών εκλογικών διαδικασιών. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε εμείς υπεύθυνοι. Εάν δεν το κάνουμε, αν δεν προστατεύσουμε την ελευθερία μας, θα είμαστε υπεύθυνοι για την επιδείνωση της δημοκρατίας στις χώρες μας και παίζεται εδώ, διακυβεύεται η αξιοπιστία μας. Ο κύριος Ραφαήλ Κλούξμαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακόμα μια φορά συζητούμε την ανάμειξη εξωτερικών δυνάμεων στις εκλογές μας. Αυτή τη φορά είναι κατόπιν αιτήματο των Άγγλων φίλων μα. Πριν ήταν κατόπιν αιτήματο των Ιταλών φίλων μα. Και αυτό θα συνεχιστεί ούτω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εναντί αυτού. Θα περάσουν πέντε χρόνια να θρυνούμε λέγοντα ότι ο Πούτιν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χειραγωγεί το εκλογικό μα σύστημα. Θα περάσουν πέντε χρόνια πολλαπλασιάζοντα τα ψηφίσματα, τα κενά και δεν θα κάνουμε τίποτα. Εμεί ε, προτείναμε μια ειδική επιτροπή επιφορτισμένη με την έρευνα αυτή τη παρέμβαση και θα πρέπει να βρει τα μέσα να το καταπολεμήσει το φαινόμενο. Και για πολιτιστικού λόγου, για πολιτικού λόγου δεν υπερψηφίσετε αυτή την επιτροπή, για πολιτικά παιχνίδια. Και αυτό θα καθυστερήσει την προσπάθειά μα. Τώρα λοιπόν, είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να σταματήσουμε να σχολιάζουμε τι εξωτερικέ παρεμβάσει και θα πρέπει να δράσουμε, να δημιουργήσουμε αυτή την ειδική επιτροπή, να κάνουμε συστάσει που προστατεύσουν τι δημοκρατίε μα. Πρέπει να δράσουμε, διότι οι αντίπαλοι μα εκείνοι δεν περιμένουν να ξυπνήσουμε για να δράσουν. Ευχαριστώ. Ναόμι Λόγγ. Ευχαριστώ. Το μέσο των γενικών εκλογών και τη εκστρατεία του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να παγρυπνούμε όσον αφορά τι απειλέ κατά των δημοκρατιών μα από ξένε εξουσίε και τουλάχιστον βλέποντα τα μαθήματα από το δημοψήφισμα του ε, Brexit. Ερευνητικοί δημοσιογράφοι αποκάλυψαν τα σκοτεινά χρήματα που έρευσαν μέσω τη Βόρεια Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία ε, την τελευταία εβδομάδα ε, του δημοψηφίσματο. Οι ακόμη σκοτεινέ όμω λεπτομέρειε δεν έχουν αποκαλυφθεί και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα δεν γνωρίζουμε το βαθμό τη ρωσική παρέμβαση στον πολιτικό μα κόσμο. Ο Μπόρι Τζόνσον αρνείται, βλέπετε, να δώσει την έκθεση των μυστικών υπηρεσιών όσον αφορά τι μυστικέ δράσει των Ρώσων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπω καταναλώνουμε τι πληροφορίε και διεξάγουμε την πολιτική μα στην ψηφιακή εποχή, είμαστε ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση και στην επίθεση ψηφιακή, είναι και εκείνου που οργανώνονται τι επιθέσει από το εξωτερικό. Τα κοινωνικά μέσα, οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δεν έχουν κάνει το σωστά. Εκείνος που διεφύβρε, ο Μπένσε που εφήβρε το διεθνές το διαδίκτυο ζήτησε να επιτεθούμε κάτι τη Αλλά και παλιά υπήρχε ένας τρόπος τη πραγματικότητας. Στη Βόρεια Ιλανδία, και υποψήφοι και τα κόμματα ήταν θύματα απειλών και πιέσεων από τους παραστατιωτικούς αυτές τι εκλογές. Θα πρέπει να εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την ακαιρεότητα της δημοκρατίας μας. Σας ευχαριστώ. Κύριος Στάνισλαφ Πόλτσακ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρέμβαση στις δημοκρατίες μας και στις ε, εκλογές μας ε, είναι απίστευτα σοβαρή ε, και αυτά τα φαινόμενα υπήρχαν και κατά το παρελθόν. Το θέμα είναι τι εργαλεία έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. Αν ήδη έχουμε χάσει κάποιες μάχες, δείτε παραδείγματος χάρη τι έγινε με το Brexit. Και θέτω το ερώτημα, μήπως αυτό πρέπει να είναι μοντέλο για μας αυτή η περίπτωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο σαν δημοκρατία έχασε αυτή τη μάχη, αλλά αυτό ίσως μας οδηγήσει να σκεφτούμε ε, μια κάποια πανευρωπαϊκή δράση. Ε, εμπιστεύομαι την Επίτροπο πάνω σε αυτό και γνωρίζουμε ότι οι αξίες της δημοκρατίας των ελευθέρων εκλογών ε, που τονίζει τακτικά πρέπει να αποστηριχθούν και ξέρουμε ότι αυτές οι αξίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είχαμε υποθέσεις ε, που ξέσπασαν και αποκαλύφθηκαν και ήταν η κορυφή του παγοβούνου, Υπάρχει παρέμβαση από Ρωσία, από Κίνα και από άλλες χώρες. Το έχουμε ακούσει. ρωσικά εργαλεία, το ρωσικό εργαλείο είναι ψέματα, ψευδείς ειδήσει, ε, παραπληροφόρηση και αποσύνθεση των ε, κοινωνιών μας από όλες τις χώρες που έχουμε αναφέρει εδώ, θα ήθελα να αναφέρω και την τσεχική δημοκρατία και την έκθεση που έχουν εκδώσει υπηρεσίες ασφαλείας. Η υπηρεσία ασφαλείας συνεπέρανε ότι η Ρωσία προσπαθεί να χειραγωγήσει διαδικασίες λήψεως αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα κυβερνήσεως, χρησιμοποιεί οικονομικά, στρατιωτικά μέσα και πιέσει σε επίπεδο ενημέρωσης και προβάλλει ατέλειες δημοκρατικών διαδικασιών. Όπω αργέ διαδικασίε, νομοθετικέ, διάφορε διοικητικέ διαδικασίε κλπ. Πιστεύω ότι με μονομένε ε, δράσει ε, δεν θα λειτουργήσουν. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα δεν αρκεί. Πανευρωπαϊκή δράση απαιτείται και αυτό πρέπει να κάνουμε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Τσίμος Τσέτσιπτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις τελευταίες παρεμβάσεις ε, στις δημοκρατικές διαδικασίες και στην ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική άλλων κρατών. Τα γνωρίζουμε αυτά από την ε, ιστορία. Είναι δυνατόν πλέον με τις νέες τεχνικές ε, να στείλει κανείς ψευδείς ειδήσει σε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς να αποκαλύπτει τους συντάκτες. Και έτσι αυτοί που λαμβάνουν τα τις ειδήσει δεν έχουν καμία δυνατότητα να ελέγξουν την ακρίβεια των ειδήσεων. Δυστυχώ θα συμβούν χειρότερα, σύντομα. Η επανάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ατελείωτες δυνατότητες ε, για να δίδονται ψευδείς ειδήσει. Ε, οι ε, άνθρωποι, οι πολίτες σε απολυταρχικά καθεστώτα ε, κινδυνεύουν πάρα πολύ. Το κοινοβούλιο αυτό έχει μια ειδική εντολή και φέρει και ευθύνη οφείλει να αποκτήσει νέα εργαλεία για να μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο που του ανήκει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος κύριος Αστραβίτσιος έχει το λόγο. κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο σπίτι της ιστορίας ε, η έκθεση ξεκινάει ε, παρουσιάζοντας την απαγωγή της Ευρώπης. Φοβάμαι ότι η σημερινή Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη με παρεμφερείς προσπάθειες. Αλλά αντί αυτού του γοητευτικού θεού βλέπουμε το διαδίκτυο το οποίο χάρη τη σύγχρονη τεχνολογία δεν χρειάζεται καν να διασχίσει φυσικά σύνορα. Οι εισβολεί υπονομεύουν τι δημοκρατικέ μα διαδικασίε και θέτουν σε κίνδυνο τις αξίες μα. Η απάντηση σε όλα αυτά θα πρέπει να είναι ο κοινό μα αγώνα για το κοινό μα μέλλον. Στη δική μου τη χώρα, τη Λιθουανία, οι δημοσιογράφοι και η κοινωνία των πολιτών ήταν οι πρώτοι και πιο αποτελεσματική στο να αποκαλύψουν ρωσική παραπληροφόρηση και να αυξήσουν την αντίσταση της κοινωνίας μας. Τον προηγούμενο μήνα περάσαμε ένα νομοσχέδιο για εκλογικές παρεμβάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει έρθει η στιγμή για να δραστηριοποιηθούμε και όλες οι σωστές προσεγγίσεις αναφέρονται στο ψήφισμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Σβέρ, ε, δύο λεπτά παρακαλώ. Σβέρ Μίλαν. Πρόεδρε, είναι πλέον πιθανό ε, να γίνουμε θύματα εκείνων που κάνουν προπαγάνδα, που καταστρέφουν την, ε, τις υποδομές ε, και διαδίδουν ψευδείς ειδήσει. Ο αριθμός των κυβερνογκλημάτων αυξάνεται και οι στόχοι δεν είναι πλέον μόνο οι κυβερνήσεις και οι πολυεθνικές, αλλά επίσης και οι οικονομικές υποδομές ε, και, τα, και απροστάτευτοι πολίτες. Οι επιτιθέμενοι κατά κανόνα δεν λειτουργούν μόνοι τους. Ο κυβερνοπόλεμος σημαίνει ότι ε, πλέον έχουμε τους εμπειρογνώμονες όπου ένας απλός ε, ιός στους υπολογιστές μπορεί να προκαλέσει μια ζημιά όπως και μια ε, στρατιωτική επίθεση. Έχουμε λοιπόν κυβερνοπόλεμο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, κατά των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ρώσοι έχουν παρέμβει στην εκστρατεία του Brexit και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Επίσης, έχουμε έγγραφα που καταδεικνύουν τις προσπάθειες του Πούτιν να ασκήσει επιρροή στις εκλογές της Ηνωμένης Πολιτείας. Αλλά εμένα δεν με ανησυχούν οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί αυτές εντόπισαν την απειλή έγκαιρα και είναι πλέον ε, ε, προστατευμένες. Ανησυχώ περισσότερο για την Ευρώπη, για την ασφάλεια των δικών μας των θεσμών. Οι απειλές αυξάνονται και σε μέγεθος και σε πολυπλοκότητα αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Φαντερ Λάιεν, γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα και σήμερα ανέφερε ότι ο νέος φορέας για την κυβερνοασφάλεια ε, θα ε, προσφέρει μια συντονισμένη Ευρώπη. Εγώ προτιμώ μια ενιαία αντίδραση, αλλά έστω και αυτό είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη η Αντιπρόεδρος ε, κυρία Ντόπρεφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι χρησιμοποιώντας ε, ε, και χειραγωγώντας τις δημοκρατίες ε, είδαν το φως οι δικτατορίες με τέλος τραγικό κάθε φορά. Και σήμερα, τον, ε, αν σκεφτούμε την ιστορία του 20ου αιώνα, η, η ιερή και όσια ελευθερία λόγου είναι αυτή που χρησιμοποιείται ακριβώς για να επιτεθούν οι κακόβουλες στη δημοκρατία. Ακριβώς αυτό προκάνει η Ρωσία. Προσπαθεί να διχάσει, να σπείρει τη διχόνοια στην Ευρώπη. Και αυτό το κάνει χρησιμοποιώντας ε, τη βοήθεια των ακραίων κομμάτων. Το βλέπουμε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αυστρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα ε, είναι ε, ότι στη χώρα μου, την Ουγγαρία, η ίδια μου κυβέρνηση το κάνει αυτό. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά. Αξιότιμε Πρόεδρε, κυρία Γιούροβα, μιλάμε για χειραγώγηση και ψευδείς ειδήσει. Ε, δεν αρκεί να υιοθετήσουμε νομοσχέδια. Χρειαζόμαστε δημοκρατικές τεχνολογίες που να είναι πιο αποτελεσματικές από τα μέσα που χρησιμοποιούν η Ρωσία και η Κίνα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υπονομεύονται οι αξίες μας. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται και στρέφεται κατά των δημοκρατιών μας. Αυτά είναι τα μέσα των εχθρών μας. Χρειαζόμαστε ακόμα πιο ευφύης τεχνολογίες για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από αυτές τις ψευδείς εκστρατείες. Για να γίνουν όμως όλα αυτά ε, χρειαζόμαστε επενδύσεις ε, κυρίως στο Horizon Europe, στην ψηφιακή Ευρώπη Χρειαζόμαστε ένα αμυντικό ταμείο της Ευρώπης και πρέπει να ε, στηρίζουμε την αλήθεια και τα σωστά μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Μπενιφέη Μπραντό. Πολλά σοβαρά επεισόδια βλέπουμε παρέμβαση με αυξανόμενη ε, συχνότητα να σημειώνονται. Έχουμε μακρύ κατάλογο από την Cambridge Analytic σε διάφορα τα δάνεια του 2016 στο Front National, η κατηγορία χρηματοδότηση παράνομη προ το κόμμα τη ελευθερία τη Αυστρία, οι δημοσιονομικέ έρευνε και κατά τη Λέγκα στην εκστρατεία για τι εκλογέ, τι ευρωεκλογέ. Πρόσφατα μάθαμε την απόφαση του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να μπλοκάρει τη δημοσίευση μιας εκθέσεως που περιμένει τα αποτελέσματα 18 μηνών ερευνών όσον αφορά ενδεχόμενη παρέμβαση των Ρώσων στην Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε το καθήκον να υπερασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολίτε μα από αυτέ τι επιθέσει που είναι μια μορφή υβριδικού πολέμου, καμιά φορά αποσταθεροποιεί την δημοκρατία μα. Χρειάζεται μια ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να ρίξει φω σε αυτά τα στοιχεία. Μη άπαξια απαντό. Ήδη ολομέλεια στι 10 Δεκεμβρίου, μεγάλη διαφορά, ψηφίσαμε σαφέ ψήφισμα που λέει ότι χρειαζόμαστε νέα μέσα. Ποιο καταψήφισε, η Λέγκα του Σαλβίνη και το Brexit Party του Φαράτζ, το Πλάνο National τη Μαρή Λεπέν. Παράξενο, ακριβώ αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Παγκαζαουρτουντούα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε Γιούροβα, χρειαζόμαστε μια ειδική επιτροπή που να ασχοληθεί με τις παρεμβάσεις και την παραπληροφόρηση για να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν εδώ και πολλά ακόμα για να υπερασπιστούμε την τη δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάποια στοιχεία. Κάποια... Η δική μας χώρα είναι θύμα της ρωσικής επέμβασης στην Καταλωνία για να αποδυναμωθεί η Ισπανία. Ε, επίσης, ιδιωτικά ρωσικά κονδύλια ε, χορηγούν διάφορα site web στα ισπανικά και διαδίδουν θέσεις ε, ακροδεξιές. Αυτή την εβδομάδα μάθαμε πως ένας κατάσκοπος της, της μονάδας ελίτ της Ρωσίας επισκέφθηκε την Ισπανία το 2006 όταν τα μέσα του Κρεμλίνου δημοσίευαν τα πρώτα ψευδή, τις πρώτες ψευδή ειδήσει όσον αφορά την ανεξαρτησία της κατασκοπής Καταλωνίας. Γιατί αποδυναμώνοντας την Ισπανία αποδυναμώνουν ολόκληρη την Ευρώπη και τη δημοκρατία μας. Γι' αυτό, Επίτροπε, πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να δημιουργήσουμε μία ειδική ερευνητική επιτροπή για αυτή την υπόθεση. Τη χρειαζόμαστε, χρειάζεται να υπερασπιστούμε τις δημοκρατίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Φαγιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε επιτυχώς κάποια μέλη για την ε, μείωση των ε, παρεμβολών και των παρεμβάσεων στις ευρωεκλογέ του 2019. Προτείνω η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή της, ε, να μελετήσει τις βέλτιστες πρακτικές και τις διάφορες τεχνολογίες που υπάρχουν και να εξετάσει τη δυνατότητα να ανατεθούν σε εθνικό επίπεδο οι αρμοδιότητες εφόσον πηγαίνουμε για πάνω από 10 εκλογές στα κράτη-μέλη μόνο τον επόμενο χρόνο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το ότι στη Ρωσία δεν μας κάνει να λησμονούμε αυτά που κάνουν άλλες χώρες. Ανησυχώ όσον αφορά την εξάρτηση Ευρωπαϊκή Ενώσεω, όσον αφορά το ξένο λογισμικό, υποδομέ και τεχνολογίε, Πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα και προσπάθεια στο να αναπτύξουμε δικό, δικά μα μέσα προστασία αν θέλουμε να παραμείνουμε μια δημοκρατία που ηγείται. Υπό το φω όλη τη παραπληροφόρηση και των ψευδών ειδήσεων, για μία ακόμη φορά απευθύνω έκκληση για συστημητική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη σημασία που έχουν τα μέσα ενημέρωση και υπεύθυνη δημοσιογραφία και στα σχολεία να γίνει αυτό και στο κοινό αυτή η ενημέρωση. Ευχαριστώ. Ο κ. Σιμέτσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω σλοβακικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε ότι οι δίκες και ελεύθερες εκλογές είναι η βάση μιας δημοκρατικής διαδικασίας και το πρόβλημα της παρέμβασης από το εξωτερικό είναι μεγάλο. Και ε, υπονομεύεται η νομιμότητα των ε, αποφάσεων που λαμβάνονται μετά τι κυβερνήσει. Δεν μιλάμε για απλέ χειραγωγήσει. Μιλάμε για το διαδίκτυο, fake news και παραπληροφόρηση, αλλά μιλάμε επίση και για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και εκστρατιών από το εξωτερικό. Και ξέρουμε διάφορε περιπτώσει από την Ευρώπη, το Βρετανικό δημοψήφισμα ή τι εθνικέ εκλογέ. Αυτό που πρέπει να γίνει και έχει συζητηθεί εκτενώς πρέπει να ενισχύσουμε τα εφιστάμενα μέσα Statcom East ή συστήματα έγκαιρης ε, προειδοποίησης και πρέπει να επενδύσουμε στην κυβερνοασφάλεια ε, ούτω ώστε να μην κινδυνεύουν οι αξίες μας που θέλουμε να προστεύσουμε. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε οτιδήποτε πρέπει να το κάνουμε μαζί. Διότι μια επίθεση επί των δημοκρατικών εκλογών σε μια χώρα σημαίνει μια επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος ε, Ματζορίνο Φραντσέσκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ζούμε σε σταθερές οικονομίες, ε, δημοκρατίες, όριμες δημοκρατίες που είναι απολύτως απαραίτητες για να έχουμε ειρήνη και το σεβασμό της αξιοπρέπειας των πολιτών. Σταθερείς και όριμες δημοκρατίες οι οποίες όμως αποδεικνύονται και ιδιαίτερα έφτραυστες, ε, δέχονται επιθέσεις, διάφορες επιθέσεις από εκστρατείες παραπληροφόρησης ε, μέχρι και από παράνομα μας χρηματοδοτήσεις και έχουμε δει και εξωτερικές παρεμβάσεις που είναι πολύ ανησυχητικές και επικίνδυνες που μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να ενταθούν. Παρεμβάσεις οι οποίες ε, ωφελούν εκείνες τις χώρες που έχουν ένα και μόνο στόχο να καταστραφεί η Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι. Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει και υπάρχουν πολλές ε, γκρίζες ζώνες, παραδείγματο χάρη αυτή την ντροπιαστική συμπεριφορά του ε, κυρίου Σαλβίνη ο οποίος ακόμα δεν είχε το πολιτικό τάρος να δηλώσει δημόσια ε, για αυτά τα περίεργα τα οποία τον συνδέουν με τη Ρωσία. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές επαφές, τις οποίες πρέπει να διαλευκάνει. Ευχαριστούμε. Ο τελευταίος ε, παρεμβαίνω είναι ο κύριος Κοβάρικ Όντρεϊ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και να, ε, ε, να ε, ευχηθώ επιτυχία για όλους σας. Ε, γνωρίζουμε όλοι μας ότι υπάρχει μια εύθραυστη κατάσταση. Πρόσφατα οι Τούρκοι ε, εόρτασαν την επέτειο της επανάστασής τους και αυτό μας το υπενθύμισε αυτό ακριβώς που σας είπα, αυτά που υπονομεύουν τις κοινωνίες μας, ε, τις ελεύθερες ανώθευτες εκλογές. Να επαγρυπνούμε σε ξένους παράγοντες που χρησιμοποιούν εκπροσώπους. Αυτό που λένε στην Επιτροπή ως κοινή απειλή. Να υπάρχει αντίσταση, να κάνουμε ένα βήμα βήμα προς την ε, καταπολέμηση εκλογικών παρεμβάσεων. Για να το πετύχουμε όμως αυτό πρέπει να επιτύχουμε την ε, ισορροπία ανάμεσα σε στοχευμένες δράσεις ε, και την προστασία της δημοκρατίας μας. Οι θεσμοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνοι τους, πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο περιβάλλον, γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα σωστά εργαλεία, να λάβουμε μέτρα κατά της παραπληροφόρησης. Να αναλάβουμε δράση για να δείξουμε εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, στις κυβερνήσεις, στα μέσα ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία και εμείς ευχαριστούμε πολύ και ε, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε πλέον αυτή τη συζήτηση. Ε, συγχαίρω την επανεκλεγήσα επίτροπο, την κυρία Γιούροβα και θα ήθελα να της δώσω και το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια που μου έδειξαν πόσο υπεύθυνοι και, και ισχυρή θα πρέπει να είμαι ειδικά για αυτό το θέμα γιατί αυτή η συζήτηση ήταν ε, πολύ ε, σημαντική και έχει υπαρξιακή σημασία για την Ένωση γιατί υπερτριγυριζόμαστε ε, από δόγματα ε, για τους οποίους όσο χειρότερα είναι η Ευρώπη τόσο καλύτερο. Ε, επίσης, 100 ε, φορές αν πεις ένα ψέμα αυτό μετατρέπεται σε αλήθεια και το ξέρουμε αυτό και από το παρελθόν, ειδικά από το τις πρώην κομμουνιστικές χώρες όπου έζησα εγώ το μισό της ζωής μου σε μια τέτοια χώρα πλήση εγκεφάλου καθημερινή γινόταν. Ε, προπαγάνδα η οποία δημιουργείται στο Κρεμλίνο και είμαι πολύ ευτυχισμένη που μπορώ εγώ να ασχοληθώ με αυτό το θέμα γιατί έχει να κάνει με ρωσική προπαγάνδα η οποία διαχέεται στην Ένωση. Ε, δεν μπορούμε μόνο όμως να κατηγορούμε τους εξωτερικούς ε, ε, φορείς, γιατί έχουμε και δικούς μας ε, σκληρά εργαζόμενους και ικανούς παραγωγούς ψευδών ειδήσεων εντός της Ένωσης. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς για το ποιους έχουμε εναντίον μας, να καταλάβουμε ποιοι είναι οι εχθροί. Πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα επηρεάστηκαν διάφορες εκλογές τα τελευταία χρόνια Προσπαθούμε να το πείσουμε το πώς και γιατί. Επίσης ε, δεν θα πρέπει να είμαστε παθητικοί, να συνεχίσουμε ε, τα όσα έχουμε ξεκινήσει, να, αναβαθμίσουμε όλες τις προσπάθειες στα σχέδια που έχουμε γύρω από τις εκλογές ε, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να συνεργαζόμαστε με τις πλατφόρμες που υπέγραψαν τον κώδικα, τον κώδικα ε, κατά της ε, παραπληροφόρησης. Επίσης, η συζήτηση δείχνει, μας έδειξε πού εξακολουθούν να υπάρχουν κενά. Εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε κατά του παράνομου περιεχομένου. Υπάρχει παράνομο περιεχόμενο που εμείς εντοπίζουμε και που ορίζουμε ως παράνομο από την νομοθεσία μας. Δηλαδή, παιδική πορνογραφία, τρομοκρατία και παράνομος λόγος μίσους που διαδίδεται. Ό,τι απαγορεύεται offline θα πρέπει να απαγορεύεται και online και θα πρέπει να ε, προβλέπετε επίσης ε, τιμωρία, ποινή. Δεν μπορεί να λειτουργεί αυτός ο χώρος ε, εκτός νόμου. Έχω συζητήσει με εισαγγελίες και πρέπει όντως να διωχθούν οι υποθέσεις παράνομου περιεχομένου online. Τώρα, για τα ψέματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παράνομο περιεχόμενο, γιατί τα ψέματα ανέκαθεν κυκλοφορούσαν ε, και δεν απαγορεύονται δια νόμου. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι αυτού του είδους τα ψεύδη και η παραπληροφόρηση ε, θα πρέπει όμως να ενεργήσουμε κατά και των υβριδικών απειλών, γιατί αυτέ συνδέονται με την ασφάλειά μας. Θα πρέπει να ε, ε, φτιάξουμε ορισμό για την παραπληροφόρηση, να εστιάσουμε σε αυτό και να εστιάσουμε και την προσοχή μας. Εργαζόμαστε για έναν ορισμό ότι αυτή η παραπλανητική ενημέρωση ε, είναι πολύ σημαντική και δημιουργεί ε, ε, προβλήματα γιατί θελημένα παραπλανεί το κοινό. Για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι δεν αγωνιζόμαστε κατά απόψεων, αλλά κατά των ψευδών ειδήσεων που είναι αποδεδειγμένα ψέματα. Και αυτά μπορούμε να τα αποδείξουμε.